Good morning everyone. Καλημέρα σε όλους. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 ε, και 7 πρώτα λεπτά να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε όλοι και περνάμε στο σημείο 6. Γενικό Επιλογισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, να σας θυμίσω ότι Έξι δημοσιονομικές ε, τροπολογίες έχουν γίνει αποδεκτές και απαριθμεί τις ε, τροπολογίες αυτές. Είναι εκτός αρμοδιότητας ε, της Επιτροπής μας, γι' αυτό δεν τις δεχτήκαμε και άλλες δύο δεν είναι αποδεκτές επειδή θεωρούνται οι προτινόμενες αλλαγές παράνομες. πριν περάσουμε την ψηφοφορία, θα δώσω το λόγο σε Μιχάλ Γκάλερ. Ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσω, σε σχέση με αυτά που υπόθηκαν χθε, ότι θα υπάρξει αυτή η προφορική τροπολογία για την τελευταία ψηφοφορία 52-57. Η τροπολογία που αφορά το επιπλέον προσωπικό σε τοπικό επίπεδο και την καλύτερη ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα εθνικά κοινοβούλια. Ε, και την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας εκεί. Εκεί ζητούμε 400.000 ευρώ περισσότερα για τις εν λόγω χώρες. Μάλιστα, ο Μιχαήλ Καλιανού εισηγητής για το θέμα αυτό, όπως γνωρίζετε. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Όχι. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας υποσχέθηκα ότι θα ψηφίζουμε αργά. Έχουμε δύο μισή χρόνια μπροστά μας για να επιταχύνουμε. Λοιπόν, όλοι έχετε την κάρτα σας φαντάζομαι, την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Πράσινο, κόκκινο και άσπρο, υπερκατά αποχές, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, 55 άτομα βρίσκονται εδώ σήμερα, αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Εντάξει, υπάρχει απαρτία. Ξεκινούμε. Πεντεπτά. 57 στους 57 υπέροχα 20, 46 ε, υπέρ 46 υπέρ κατά αποχές 5347, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. ηλεκτρονική ψηφοφορία ε, τη γνωρίζετε, όσοι ε, αλλιώ την ανατενάση χειρό. 53-37 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 53-35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-04 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. Το 53, 5305 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5306 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε τώρα 53, 26, 25, 26, 27. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53, 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53, 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 53-54 υπέρ. Κατά αποχές θα πρέπει να το ελέγξουμε αυτό. 53-54 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. The vote is... Πέρας ψηφοφορίας. Καλή αρχή, μάλιστα. Απορρίπτεται. 53-17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές Ας τον ελέγξουμε το συμβασμό 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα is Δεν χρειάζεται να το τσεκάρουμε τελικά. Συμβασμό 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5315 53-15. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5319 53-19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 5320 53-20. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 53-58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 53-29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-21 υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε το 53-21 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. 53-21 τροπολογία του κ. Πάετ και άλλων. Λοιπόν, ακόμα πέντε συνάδελφοι, τέσσερις. Τρεις, δύο. Εν πάση πέρα πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 53-59 υπέρ, κατά, αποχές. Να το ελέγξουμε το 53-59, την τροπολογία Γκίλ, άρχιτη ψηφοφορία, Πέρας ψηφοφορίας. Τώρα εδώ περισσεύει κάποιος το ΕΛΚ. Απορρίπτεται. Και 53-22 υπέρ. Κατά αποχές. δύσκολο να συζητήσουμε και καινούργια σύνθεση γενικά εδώ. Να το ελέγξουμε παρακαλώ το 5322. Ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Κοιτάζαμε τι κάνουν οι φιλελεύθεροι και ξέραμε τι γίνεται. Αλλά δεν είναι πια έτσι τα πράγματα. Δεν σας λένε καν φιλελεύθερους, μάλιστα. Κοιμούνται έξι συνάδελφοι ακόμα. Ωραία. Ε, εντάξει. Πέρας εγκρίνεται 5360 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5223 53-23 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ομαδική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5301 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5376 Καστάλντο υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται. 5363 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5364 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβασμός 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβασμός 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52-62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53-72 υπέρ κατά αποχές 53-72 θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 5373 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5374 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εδώ δεν ψηφίζουμε. Μεγάλη μαθητική ψηφοφορία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν έχουμε τελική ψηφοφορία από ό,τι μου λένε. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε λοιπόν. So after our spectacular voting... Λοιπόν, μετά την εντυπωσιακή αυτή ψηφοφορία που είχαμε, θέλουμε να συνεχίσουμε τώρα. Και περνάμε στο σημείο 11. Ανταλλάξαμε το 7 και το 11 τη σειρά του. Ενημέρωση σχετικά με τι βουλευτικέ εκλογέ στην Ουκρανία που έγιναν στι 22 Ιουλίου του 2019. Για τις εκλογές αυτές το Ευρωκοινοβούλιο έστειλε μια αντιπροσωπεία παρατηρητών. Εγώ είχα την τιμή να είμαι επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας και μαζί με την ε, συνάδελφο Κανιέτα, την ε, Σάντας από, την, από τους ε, σοσιαλιστές, τον κύριο Αστρολίσο, την Γιούλια Βαν από τους Πράσινους, ε, εκπροσώπους από το ECR και από το EFD. Παρατηρήσαμε αυτές τις εκλογές, ήμασταν παρατηρητές μόνο σε αυτές τις εκλογές στην πόλη του Κιέβου. Δεν είχαμε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε σχετικά με το έργο μας και το αποτέλεσμα των εκλογών, οπότε θα το συζητήσουμε σήμερα εν συντομία το θέμα αυτό. Θυμάστε, ε, ε, πρόκειτο για πρόορες εκλογές μετά τη διάλυση του Κοινοβουλίου από τον ε, νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ζελένσκι στα τέλη του Μαΐου, κάτι που έγινε ω πρώτο μέτρο την μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Το Ευρωκοινοβούλιο ε, συμμετείχε ως παρατηρητές. Παρατηρητές έστειλαν και άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Οι εκλογές έγιναν ομαλά, ε, με σεβασμό των θεμελιωδών ε, ελευθεριών, αν και υπήρξαν κάποια προβλήματα ε, με σύγκρουση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων, κάποιες ελλείψεις και στην ελευθεροτυπία. Να Πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εκλογές αυτές έγιναν στο πλαίσιο της ε, ρωσικής επιθετικότητας ενάντια, τη... ενάντια στην ε, Ουκρανία, μενόμενης ακόμα της, ε, της έντασης που υπάρχει στην Κρυμαία και στον Ντονμπάς. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι οι εκλογές δεν έγιναν στην Κρυμαία, εδάφη που ε, ελέγχονται επίσης παράνομα από στρατεύματα στο Ντομπάς και οι 26 έδρες που ανήκουν σε αυτές τις περιφέρειες παραμένουν κενές. 49% ήταν συμμετοχή, 5 κόμματα ε, υπερέβησαν το κατέφυλλο του 5%, η πρωτοβουλία για τη ζωή, το κόμμα ε, για την πατρίδα, η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη, το κόμμα του πρώην Πρόεδρου Πορσένκο και τέλος το Κολός. Οι εκλογές ε, επέφεραν μεγάλη αλλαγή στη σύνθεση του Κοινοβουλίου με το κόμμα του κ. Ζεντένσκι, το οποίο ιδρύθηκε μόλις πριν από λίγους μήνες και δεν εκπροσωπούνταν στο προηγούμενο ε, κοινοβούλιο, α, κατέλαβε πλέον 2,54 έδρες από τις 450. Πρόκειται επίσης για ένα πολύ νέο ε, κοινοβούλιο. 68% ε, των ε, βουλευτών ε, έχουν ε, ηλικία κάτω των 45-46 ετών. Η Ουκρανία, όπως έχουμε συζητήσει πολλές φορές, ε, παραμένει στενός και στρατηγικός σύμμαχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη συνδράμουμε στρατηγικά και με κάθε πρόσφορο μέσο. τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα πρωτοφανέ επίπεδο συνεργασία ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, την, το Κοινοβούλιο τη ε, Ουκρανία, με διάφορου διαλόγου, ακόμη και μεταξύ πολιτικών κομμάτων και πολιτικών ομάδων. Στο πνεύμα λοιπόν του διαλόγου και του συμβασμού, ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επέμεινε στην ανάγκη να υπάρξει κλίμα συνένεσης στο νέο Κοινοβούλιο. Και ε, προσβλέπουμε στην ε, καλή συνεργασία μελλοντική με την Κοβναράντα, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, με τον Πρόεδρο ε, ιδίω και ο αντιπρόεδρος, ε, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, πραγματοποίησε και επίσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα στο, Ευρωπαϊκό, στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας στο πλαίσιο αυτών των νέων σχέσεων που θέλουμε να δημιουργήσουμε. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στα μέλη αυτής της αντιπροσωπής αν τα κανιέται. Ευχαριστώ. Ήταν πραγματικά ε, συγκινητικό το να είναι κανείς παρατηρητής σε αυτές τις εκλογές. Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν και κάποιες παρατυπίες στην εκλογική διαδικασία, μπορούμε να πούμε ότι οι εκλογές αυτές διεξήχθησαν ομαλά, ήταν δημοκρατικές εκλογές και τα πιο σημαντικά πράγματα που είδα εγώ ω εικόνε ήταν η κατάσταση στην ε, Λευκορωσία, η κατάσταση στην Ουκρανία και στη Ρωσία. Στη Ρωσία εδώ και πάνω από 20 χρόνια ε, στην ουσία έχουμε δύο φάσεις. Μετβέντεβ ή Πούτιν. Πούτιν. Στη Λευκορωσία Μετβέντεβ, ε, Λουκασέγκο και στην ε, Ουκρανία υπάρχει ε, μια παρόμοια κατάσταση. Αυτό που θέλω να πω δεν είναι για τις εκλογές. Έχουν αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργούς στην Ουκρανία. Θέλω να πω ότι η επικεφαλής των σχέσεων μας με την Ουκρανία θα είναι ο πολύ έμπειρο. ε, κύριος Τζιντζάτσε. Όμως πρέπει να αλλάξουμε και τη στάση μας απέναντι στην Ουκρανία. Ε, ιδίως όσον αφορά τον, ε, τον, την, ε, τον ύπατο εκπρόσωπο αντιπρόεδρο της ε, Κομισιόν. Η Μογκερίνη επισκέφθηκε μία, άντε το πολύ δύο φορές στη θητεία της στην Ουκρανία. Ε, επόμενο ύπατο εκπρόσωπο. αν βεβαίω επιβεβαιωθεί στη θέση αυτή από το Κοινοβούλιο, πρέπει να θέσει την Ουκρανία στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων του, διότι η Ουκρανία είναι ζωτικός, ε, ζωτικής σημασίας εταίρος για την Ευρώπη και λόγω και του γεγονότος ότι έχουμε και έχει και άλλους γείτονες που δεν είναι δημοκρατικές ε, χώρες, που δείχνουν επιθετικότητα και προσπαθούν να διχάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα ιδιωτελή συμφέροντά τους. Αυτή είναι η ευχή που θέλω να εκφράσω για τον επόμενο υπό το εκπρόσωπο και νομίζω ότι η Επιτροπή μας θα πρέπει ρητός και κατηγορηματικός να το εξηγήσει αυτό και το πόσο σημαντικά είναι για εμάς τα αιτήματα αυτά. Ευχαριστώ τη Σανδρακανιέτε. Κυρία Σάντος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Οι εκλογές ε, έγιναν ε, με συνταγμένο τρόπο και μπορούσαν να εκφραστούν πραγματικά οι πολιτικές επιλογές ε, του πληθυσμού. Αυτός ήταν, και αυτός ήταν και ο, ο πυρήνας ε, της ε, αποστολής μας. Βεβαίως είχαμε κάποιες αλλαγές στον εκλογικό νόμο, κάποιες τροποποιήσεις είναι απαραίτητες. Επίσης χρειάζεται μια καλύτερη διαχείριση σε ό,τι αφορά τελικά ποιοι είναι οι πόροι κρατικοί και ποιοι είναι οι πόροι των κομμάτων ε, οικονομική εννοώ. Από εκεί και πέρα ήταν καλό το κλίμα και η επιλογή των πολιτών έγινε ελεύθερα. Αυτό είναι και το πλέον σημαντικό. Τα υπόλοιπα προβλήματα τώρα που υπάρχουν εκεί, στην Ουκρανία, ε, στην Κρυμαία, συγγνώμη, και τον Ντομπάς, ε, και το μέλλον της χώρας ε, είναι μια άλλη συζήτηση. Είναι πολλά τα ανοιχτά θέματα. Θα γίνει και μια ακρόαση σήμερα όπου θα συζητήσουμε και άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα για το μέλλον της χώρας αυτής και για το μέλλον της περιοχής, της ευρύτερη περιοχής και της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ εγώ και τώρα από τη Renew Europe, Πέτρας. Ευχαριστώ και βεβαίως πρέπει όλοι να σας συγχαρούμε και για την πρόσφατη εκλογή σου, Γκρέαμ με πολύ καλή οργάνωση, τακτική, διεξαγωγή, έχοντας ε, παρατηρήσει εκλογές με τον συνάδελφο και στο παρελθόν στο ΒΙΦ. Διαπιστώνουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο πατριωτισμού και συναισθημάτων πατριωτικών που εκφράστηκαν. Βέβαια πάντα η Δυτική Ουκρανία είχε διαφορά από την υπόλοιπη χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως, ε, τώρα το καινούριο στοιχείο είναι ότι πριν ανοίξουν τα εκλογικά τμήματα, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο. Ασυνήθιστο για μας. Αλλά πάλι δείχνει το πνεύμα που επικρατεί. Και επίσης σημειώνεται ένα υψηλό ε, ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Η οργάνωση ήταν πολύ καλή. Μπορεί να λείπαν ένα-δύο πράγματα, λεπτομέρειες όμως, τίποτε το σημαντικό. Η Ουκρανία θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να εστιαστεί και συμφωνώ σε αυτό, Ελίζαμπετ, θα πρέπει να εστίσουμε και την υποστήριξή τους, την υποστήριξη μας, ε, να τους υποστηρίξουμε στην οργάνωση του οικονομικού σκέλους της περιοκλογικής εκστρατείας, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα διαφθοράς, να επικρατεί περισσότερη διαφάνεια. Και πάλι, όπως είπα, η Δυτική Ουκρανία διαφοροποιείται από την υπόλοιπη, καθώς ο Ποροσέγκο κέρδισε τις εκλογές, ο πρώην πρόεδρος ε, με το κόμμα του, που ηγήθηκε στα υπόλοιπα ε, της χώρας. Ήταν πολύ καλός ο συντονισμός και η εξαγωγή οργάνωση των εκλογών η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία είχε επιτυχές έργο με τις συναντήσεις της, ε, περισσότερες συναντήσεις και επαφές από ό,τι συνήθως. Αυτά και προσβλέπουμε σε πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ Πέτρας, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω. Ήταν ε, πολύ καλή οργάνωση και της ε, ευρωπαϊκής πλευράς. Βέβαια είχαμε και την μεικτή αυτή αποστολή, έτσι. Ήταν συνάδελφοι και από τον από την ΟΑΣΕ, πράγμα το οποίο διευκολύνει πολύ καθώς η κατάσταση στην, ε, σε σχέση με την Ουκρανία είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε σχέση με μία χώρα και δεν εννοώ βέβαια την Πορτογαλία, μέλος της ΟΑΣΕ. Ναι, ευχαριστώ και εγώ θα συμφωνήσω με τα όσα υπόθηκαν ε, για την οργάνωση, τη διεξαγωγή των εκλογών. Ήταν πολύ επιτυχής. Πέμπτη αποστολή παρατήρησης για μένα, η καλύτερη όχι μόνο σε όρους οργάνωσης, αλλά και σε όρους πλουραλισμού, δημοκρατικής ε, συμπεριφοράς, πνεύματος. Ήμασταν στην Οδέσα, στην, Ο... στην Οδυσσό, στην Νότια Ουκρανία και σε συνθήκες μάλλον ε, ή κλίμα μάλλον δύσκολο ως προς τις δημοκρατικές ε, λειτουργίες, αλλά τα πράγματα πήγανε καλά και ήμασταν γενικά ικανοποιημένοι όλοι. Θα ήθελα ωστόσο να εστιάσω την προσοχή μου στην κατάσταση που επικρατεί στο νεοσυσταθέν κοινοβούλιο, στο υποσύσταση κοινοβούλιο, γιατί αυτό που βλέπουμε τώρα μετά τη σύσταση του κοινοβουλίου ε, την προηγούμενη Δευτέρα, η κατάσταση δεν είναι μόνο θετική, δηλαδή ε, όταν έρθει η ώρα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής αντιπροσωπή σε μερικές ώρες, θα ήθελα να σταθούμε και στη συμπεριφορά του νέου Προέδρου όπως και της νέας κυβέρνησης, διότι δεν είναι εύκολο να διαγνώσει κανείς να προβλέψει τι θα προκύψει σε αυτή την κατάσταση. Όπως είπε και ο Ντέβιτ Μακάλιστερ, έχουμε ένα περίπου 80% των βουλευτών εκλεγέντες βουλευτές χωρίς προηγούμενη εμπειρία από κοινοβουλευτικό βίο και μάλιστα χωρίς πολιτικό πρόγραμμα χωρίς δομές, χωρίς ε, μια, ένα όραμα, μια ιδέα για το πώς θα προχωρήσει αυτή η χώρα. Έτσι λοιπόν, θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς ενδεχόμενα ε, αυταρχική συμπεριφορά του Σελένσκη και της κυβέρνησής του. Έτσι ώστε να μην υπάρξει μια αρνητική, ένας αρνητικός αντίκτυπος μετά την διαξαγωγή των εκλογών ε, σε σχέση με τον πρόεδρο και την κυβέρνησή του. Βεβαίως ξέρω ότι όπως πες και εσύ έχουμε πολύ ικανούς ε, ανθρώπους στην Ουκρανία, ωστόσο εμείς οι Ευρωπαίοι αλλά και ε, η αντιπροσωπεία με το η νέα της ηγεσία πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις. Ο κ. Σελένσκι δεν έχει ουσιαστικά δεσμευθεί στην τήρηση της διαδικασίας για την αποκέντρωση και την μεταρρύθμιση του τομέα της δημόσιας υγείας. Τομείς ο οποίο εμείς πρέπει να σταθούμε ως αντιπροσωπεία. Μάλιστα θα πρέπει να δώσουμε ε, ιδιαίτερη προσοχή ώστε να τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις ή να υλοποιηθούν αυτές οι μεταρρυθμίσεις καλύτερα και να υποστηρίξουμε το Σελενσκή στην ε, εισαγωγή νέων μεταρρυθμίσεων που θεωρώ απαραίτητες. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ιντε, ο κύριος Μπέρκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και πολύ σύντομα. Καθώς οι συνάδελφοι έχουν ήδη πει πολύ σημαντικά πράγματα για την αποστολή αυτή, ε, σε δύο σημεία θα ήθελα να αναφερθώ, ε, γιατί ήμασταν με τον κύριο Στραβίτσιος και με την κυρία Φονπέρκ στην ε, Δυτική Ουκρανία, όπου παρατήρησα ότι οι νέοι ιδιαίτερα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό έλαβαν μέρος ε, στην εκλογική αναμέτρηση. Ε, ιδιαίτερο μέλημα βεβαίως είναι πάντα και κύριο θέμα των εκλογών είναι η εδαφική ακαιρεότητα αλλά και η διαφθορά έχει πολύ μεγάλη προβολή ως ε, θέμα στις εκλογές. Οι νέοι ιδιαίτερα μας ε, απίφθηναν το μήνυμα παγίως να μην τους εγκαταλείψουμε, να μην τους λησμονήσουμε. Αυτό εμένα με ε, εντυπωσίασε πολύ και δεν θα το λησμονήσω, θα είναι πάντα γνώμονα στις δράσεις μου και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να ευχαριστώ του συναδέλφου για την πολύ καλή συναδελφική στάση και συνεργασία στη διάρκεια αυτή τη αποστολή στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπέρκ. Αυτή ήταν η συνάδελφοι λοιπόν που έχοντας επισκεφτεί την Ουκρανία έλαβαν το λόγο. Ε, τώρα παρακαλώ τους λοιπούς συναδέλφους αν έχουν κάποια σχόλια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εγώ δεν συμμετείχα στην αποστολή, αλλά βεβαίως παρακολούθησα τις εκλογές ε, στην Ουκρανία και την εξελίξει μετά τις εκλογές. Ε, τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Ανοίγουν ε, ένα νέο κύκλο με νέες ευκαιρίες και νέες προκλήσεις. Από την εμπειρία μας, όμως Λιθουανούς, από της Βαλτικής, ε, μου θυμίζει τις πρώτες εκλογές το 1992-1993 στην ε, Λιθουανία μετά την Επανάσταση. Αυτοί που ζήτησαν την εξαρτησία της Λιθουανίας ε, και που έκαναν την επανάσταση στην πραγματικότητα έχασαν τις εκλογές. Δεν είναι βέβαια το ίδιο ακριβώς στην Ουκρανία, αλλά μοιάζει. Ο κόσμος ζητάει από τις αρχές γρήγορες αλλαγές και αυτές οι αλλαγές δεν γίνονται. Ε, δεν λαμβάνουν χώρα και ο Ποροσέγκο ήταν θύμα αυτής της ε, χαμένης προσδοκίας. Από την, όλα, από την άλλη οι αλλαγές ε, δεν αλλάζουν το 1996 άλλαξε πάλι η κυβέρνηση στη Λιθουανία. Το ίδιο θα γίνει και στην Ουκρανία και εκεί θα έχουμε νέες αλλαγές. Το που ήταν σημαντικό για μας σε όλες αυτές τις αλλαγές τις κυβερνητικές είναι ότι είχαμε πάντα κατά νου ότι πρέπει να λάβουμε χώρο μεταρρυθμίσεις. Γιατί, γιατί, γιατί υπήρχε ένα καρότο. Το καρότο ήταν η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη. Πρέπει λοιπόν να δούμε με την Ουκρανία τι συμβαίνει. Μια χώρα που είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, που είναι προκλήσει πολύ μεγάλε. Και για να μπορεί να έχουν κίνητρα για μεταρρυθμίσει οι Ουκρανοί, παρά τον ενθουσιασμό του Ζελέσνη, μπορεί και να παρά είναι ενθουσιώδη κατά κάποιο τρόπο, δεν θα είναι εύκολο. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Μπορεί σε δύο χρόνια η δημοτικότητα του κυρίου Ζελέσνη και του κόμματο του μπορεί να μειωθεί σημαντικά. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε εμεί τώρα για να βοηθήσουμε του Ουκρανού να εξακολουθούν να έχουν κίνητρα για μεταρρυθμίσει. Και από ανθρώπου υψηλό υψηλά ιστάμενου, ε, πολλοί λένε ότι ενδεχομένω πρέπει ε, να ε, επιβραδύνουμε ε, της, ε, τη διαδικασία σύγκλησης, διότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι επώδυνες, Θέλει προσοχή λοιπόν. Ας, ας μάθουμε από τις εμπειρίες μας και να είμαστε προσεκτικοί όταν ε, εξετάζουμε τι περιμένει την Ουκρανία στο μέλλον. Ο κύριος Κλούξμαν από, τους, από το S&D παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Ακούστε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, στην Ουκρανία να έχουμε ένα success story. Μιλάμε για μια χώρα που είναι ε, σε πόλεμο ουσιαστικά και που μέρος της οποίας είναι υποκατοχή. Ε, θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σαφείς και να το πούμε και στην ε, είπατε εκπρόσωπο, θέλουμε μεγαλύτερη εμπλοκή δική μας στην Ουκρανία. Διότι εάν τη βγάλουμε την ατζέντα μας θα είναι καταστροφικό αυτό και για την Ουκρανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένας τρόπος που έχουμε για να βοηθήσουμε τη νέα πλειοψηφία, τη νέα κυβέρνηση στην Ουκρανία και το λαό της Ουκρανίας είναι να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε γιατί, γιατί έχουμε επιβάλει τις κυρώσεις ε, στη Ρωσία, στον, ε, στη γειτονική χώρα. Έτσι λοιπόν στο Συμβούλιο τη Ευρώπης αυτή τη στιγμή επιστρέφει η Ρωσία και η ρωσική αντιπροσωπεία χωρίς να υπάρχει, υπάρξει καμία πρόοδο στην Ουκρανία ε, την κατοχή ε, και την ε, προσχώρηση της Κρυμαίας στη Ρωσία. Ε, δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάμε. Δεν, είμαστε, δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, έτσι. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε τον Πούτιν, έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία και να στεφτούν από επιτυχία. Και ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Ουκρανικό λαό είναι το θέμα της διαφθοράς. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε και να πιέσουμε ε, και αν θέλετε και τη νέα κυβέρνηση έτσι ώστε επιτέλους να γίνει κάτι για να μπει τέλος αυτό το μεταολιγαρχικό σύστημα που εξακολουθεί να ισχύει και εκεί. Ευχαριστώ τον κύριο Γκλούξμαν ή κάποια νάουτα. Ο κύριος, κάποια ο κύριος Νάρτ μάλλον. Ε, έχει το λόγο. Πρέπει να καταλάβουμε γιατί έλαβε χώρα αυτό το τσουνάμι στην Ουκρανία. Γιατί 80% νέοι βουλευτές ε, μπήκαν στη ράντα στο κοινοβούλιο δηλαδή της ε, Ουκρανίας και γιατί ένας ε, κομικός, ένας άνθρωπος της τηλεόρασης, ένας άνθρωπος χωρίς πολιτικό παρελθόν ήρθε και θριάμβευσε επί των παλαιών πολιτικών του Ποροσέγκο ή άλλων υποψηφίων όπως η κυρία Τιμοσέγκο. Ο κόσμος βαρέθηκε στην Ουκρανία, βαρέθηκε τους ολιγάρχες τους διεφθαρμένους, ένα εξαιρετικά διεφθαρμένο σύστημα. Έτσι λοιπόν το βασικό στοιχείο είναι ότι έχουμε ένα πληθυσμό ο οποίος υπέφερε από την διαφθορά των ολιγαρχών τους και έχει μια νέα ελπίδα απέναντι στους νέους αυτούς κυβ... κυβερνήτες. Το πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για δεκαετίες υποστήριξε αυτούς τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Έτσι λοιπόν ο λαός της Ουκρανίας, ο κόσμος, ο απλός κόσμος, που είναι αυτοί που υποφέρουν από τη διαφθορά αυτή, βλέπουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έως τώρα υποστήριζε τους διεφθαρμένους πολιτικούς. Αυτό είναι που με ανησυχεί εμένα. Σιγά σιγά υπάρχει ένα σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το είδαμε και στην Μολδαβία αυτό και η Μολδαβία ήταν θύμα ε, διεφθαρμένων πολιτικών που υποστήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να, έχουμε κατά νου ότι συμβαίνει αυτό και να είμαστε πιο κοντά στους πολίτες και όχι στους ολιγάρχες των χωρών αυτών. Thank you. Javier. Ευχαριστώ, Χαβιέρ. Ήταν ο Χαβιέρ Νάρτ. Και τώρα ο κ. Μαριανή έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, βεβαίως ε, και μπορούμε να χαρούμε που ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκλογική διαδικασία στην Ουκρανία και στις προεδρικές εκλογές, στην προεδρική εκλογή και στις βουλευτικέ. Από εκεί πέρα όμως, και συμφωνώ λίγο και με τον προηγούμενο μιλητή, πέρα από το τεχνικό ζήτημα, αλλά στο θέμα της ευρωπαϊκής, της, μάλλον της πολιτικής επιλογής, είναι ένα χαστούκι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε ε, πάση θυσία τον πρόεδρο Ποροσέγκο την πλειοψηφία του, έτσι. Χρηματοδοτήσαμε την κυβέρνηση αυτή, ενώ γνωρίζαμε ότι η διαφθορά είχε φτάσει σε ένα επίπεδο παρεμφερές με την προηγούμενη κυβέρνηση και ότι σιγά σιγά ο Ουκρανικός λαός ε, είχε τελείως χάσει ε, είχε τελείω ε, αποσύρει εν πάση περιπτώσει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση αυτή. Ε, τώρα ελπίζω η νέα κυβέρνηση να ακολουθήσει μια νέα πολιτική. Εμεί το 2015 είμαστε κατά τη συμφωνία σύνδεση με την Ουκρανία. Με ανησυχία ακούσαμε τον νέο πρόεδρο, τον κύριο Ζελίνσκι, να αναφέρεται στην, ε, το ενδεχόμενο ενό δημοψηφίσματο για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό ήταν καταστροφικό και μπορεί το σύνολο τη Υπήρου, τη Ευρωπαϊκή, να οδηγηθεί σε μια αντιπαράθεση ακόμα πιο έντονη με τη Ρωσία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς συμφωνούμε με την ε, συμφωνία του Μίνσκ. Η, συμφωνία, η συνάντηση του Σεπτεμβρίου με βάση ε, την σύνθεση της Νορμανδίας να οδηγήσει ε, σε μια συμφωνία που να είναι αποδεκτή από όλου. Έχουν πεθάνει 13.000 άνθρωποι στα ανατολικά της Ουκρανίας και από τις δύο πλευρές πλέον της εμπόλεμης ζώνης αυτής θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια για να υπάρξει κατευνασμός, ειρήνευση και όχι να υποστηρίζουμε μόνο τη μία πλευρά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαριανή. Η κυρία Ιάννα τώρα για το ECR. Thank you, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να συγχαρούμε την Ουκρανία για την ε, ειρηνική, δημοκρατική, έφτακτη μετάβαση της εξουσίας. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι δείγμα της, του εκδημοκρατισμού της χώρας παρά τις δυσκολίες και τις αντικσοότητες που βεβαίως παραμένουν αναλύωτες και τις οποίες βεβαίως θα πρέπει να τις συζητήσουμε ε, και να μην τις ξεχνάμε. Η Κρυμαία ε, εξακολουθεί να βρίσκεται υποκατοχή από τη Ρωσική Ομοσπονδία κάτι το οποίο βεβαίως εμείς δεν έχουμε κάνει αποδεκτό και έχουμε καταδικάσει. Η σύγκρουση συνεχίζεται στην Ανατολική Ουκρανία. με απλούς Ουκρανούς πολίτες να εξαφανίζονται, με πολιτικούς κρατούμενους και παρά την ε, προθυμία ε, του κύριου Ζελένσκι, η στάση της ε, Ρωσίας έχει μείνει αμετάβλητη. Θέλω να συνεχίσω βάσει αυτών που είπε η Σάνδρα Κανιέτε. Είναι μια κρίσιμη στιγμή, αυτή που διανύουμε τώρα, να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση ε, στη Ρωσία, να υποστηρίζουμε την Ουκρανική κυβέρνηση, να ενισχύουμε και να βοηθούμε στις διαδικασίες μεταρρύθμισης και να εξομαλύνουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι απλοί πολίτες της Ουκρανίας, να συνεχίσουμε να πιέζουμε για την απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων και των εχμαλώτων πολέμου. Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις ε, μειονότητες στην ε, Κρυμαία, ιδέα στους Τατάρους της Κρυμαίας. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση. Ναι, η σύνθεση του νέου Ουκρανικού Κοινοβουλίου ε, είναι ενδιαφέρουσα. Φαίνεται ότι υπάρχει μια νέα γενιά η οποία αναλαμβάνει τα ενία της εξουσίας. Συμφωνώ ταυτόχρονα βεβαίως ότι η έλλειψη ε, εμπειρίας ενδέχεται να δημιουργήσει και ορισμένα προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, θα είναι πιο εύκολο για τον πρόεδρο και την κυβέρνηση να προχωρήσουν τις μεταρρυθμίσεις, ακριβώς γιατί έχουν ε, ε, ισχυρή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και πρέπει να τους το υπενθυμίσουμε αυτό στους ε, Ουκρανούς εταίρους μας, ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα προσχήματα ε, για να ε, παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Ε, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τον διορισμό του νέου εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει λοιπόν να πιέσουμε την Φεντερίκα Μογκερίνη να αναλάβει ε, περισσότερες πρωτοβουλίες με την ε, Ουκρανία πρέπει πραγματικά να υπάρξουν συχνές επισκέψεις και δραστηριοποίηση πραγματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε Άννα Φωτίγκα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Παπαδάκη. Ευχαριστώ. Ε, συζητάμε για την υπεραλιστική επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μαϊντάν και τι είδους δημοκρατία άφησε πίσω της. Κάτι συμβολίζει ότι επικράτησε τελικά κομικός στις συγκεκριμένε εκλογέ. Οι ολιγάρχες παλιότερα είναι παλιά τέχνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ τι ακούσαμε, συγχαρητήρια, σεβασμός στην ελευθερία, πλουραλισμός. Ακούστηκε κιόλας ότι είναι και υψηλό ποσοστό το 49% και κάποια μισόλογα για ορισμένες παρατυπίες ή μήπω εννοείται μεταρρυθμίσει όπω ακούστηκε το γεγονό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα απαγορεύτηκε στι 16 του Ιουλίου από το Συνταγματικό Δικαστήριο ή και μετά από λίγο και η εφημερίδα του ανακλήθηκε η κυκλοφορία της. Το θέμα είναι το εξή, ξεκάθαρα. Θα καταδικάσετε ονομαστικά στην έκθεση που θα, θα συντάξετε τη μη συμμετοχή του Κομμουνιστικού κόμματο και την απαγόρευσή του από τη συμμετοχή στι εκλογέ ή θα επιβραβεύσετε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση συνεχίζοντας τα παχυλά κονδύλια με βάση τη συμφωνία σύνδεση που έχετε υπογράψει. Thank you, Mr. Ευχαριστούμε κύριε Παπαδάκη. Κύριε Μπότσκο. Thank you very much for the floor. Ευχαριστώ πολύ Συμφωνώ με ορισμένου από του προλαλήσαντε. θα ήθελα όμως να τονίσω ιδίως ε, τις ιδιαιτερότητες των εκλογών στην υπερκαρπασία ε, αναφέρονται και στην έκθεση ε, το γεγονό ότι το Σύνταγμα ε, εξασφαλίζει τις ελευθερίες όλων των πολιτών, ε, την ισότητα. Αυτό όμως δεν το είδαμε στην πράξη. Ιδίω στις μονοέδρικες περιφέρειες που δημιουργήθηκαν. Φυσικά προβλέπει ο νόμος ότι εκεί όπου ζουν οι εθνικές μειονότητες ε, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να ψηφίζουν σε μονοετρικές περιφέρειες για να έχουν οι μειονότητες, οι υποψήφοι των μειονοτικοί τη δυνατότητα να εκλεγούν στην, στο Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, αλλά δυστυχώς όπως και το 2014 και φέτος η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή αρνήθηκε να δημιουργήσει τέτοιες μονοεδρικές περιφέρειες και όλη η επικράτεια στην οποία ζουν οι ε, Ούγγροι από την Ουγγρική μειονότητα, άνθρωποι από την Ουγγρική μειονότητα, χωρίστηκαν σε τρεις εκλογικές περιφέρειες και έτσι δεν ε, κατάφεραν να εκλέξουν εκπρόσωπό τους. Ήταν προφανές ότι έτσι όπως δημιουργήθηκαν οι εκλογικές περιφέρειες δεν είχε τη δυνατότητα κανένας Ούγγρος μειονοτικός να εκλεγεί. Παρά το γεγονό ότι στι περιφέρειε αυτέ ε, ο πληθυσμό τη μειονότητα ανέρχεται στο 30%. Δυστυχώ ε, δεν κατέστη δυνατό ε, άνθρωπο από τη μειονότητα να εκλεγεί, από την ουγγρική μειονότητα. Γι' αυτό και θέλω να επιστήσω για άλλη μια φορά την προσοχή σα ότι τα δικαιώματα αυτά υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, στο Σύνταγμα και δεν προστατεύονται, δεν εφαρμόζονται. Πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να ασχίσουμε πίεση στην Ουκρανία να εφαρμόζει τους ίδιους τους, τους νόμους και το ίδιο της το Σύνταγμα. Είπατε ότι υπήρξαν κάποιες παρατυπίες, ε, τέτοιες έγιναν και στο, στο ε, στις περιοχές στις οποίες ανέφερα. Υπήρχαν διπλο υποψηφιότητες, υπήρχαν ε, ε, διπλή εκλογική κατάλογη, άνθρωποι που διπλοψηφίσαν, έγιναν αστυνομικές επιχειρήσεις εναντίον ακτιβιστών που συμμετείχαν στο πλευρό των Ούγγρων υποψηφίων από την μειονότητα. Ελπίζω και περιμένω ότι αυτές οι υποθέσεις ε, θα διαλευκανθούν ε, και με την συνδρομή των αστυνομικών αρχών, αν και δεν έχω και πολύ μεγάλες ελπίδες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Τσεμοτσέβιτς. Ευχαριστώ. Ασχολούμαι με τα θέματα της Ουκρανίας, με Ουκρανούς ηγέτες έχω επαφές τα τελευταία 20 χρόνια, 25 χρόνια και πρέπει να πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι η λιγότερο, η καινούρια κυβέρνηση είναι η λιγότερο προβλέψιμη από όλες τις εποχές. Διαπιστώνεται πολύ ψηλό επίπεδο κόπωσης και δυσφορίας των πολιτών που έχουν πια κουραστεί από κακές συνθήκες διαβίωσης, διαφθορά, ε, έντονη παρέμβαση και επιρροή των ολιγαρχών κτλ. Είναι δύσκολο βέβαια να προβλέψουμε τι μπορούμε να περιμένουμε από τον κύριο Ζελένσκι και την κυβέρνησή του. Πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός πως έχουν λάβει πολιτική εντολή από την ισχυρή πλειονότητα των Ουκρανών πολιτών. Αυτή είναι η εταίρη μας, με αυτούς πρέπει να συνεργαστούμε. Διαβάζοντας τα βιογραφικά μελών του, ναι, της νέας κυβέρνησης, βλέπω ότι κάποιοι είναι ε, νέοι, με καλή μόρφωση, βέβαια δεν έχουν εμπειρία. Ίσως κανείς θεωρήσει ότι μπορεί και να κάνουν μια καλή προσπάθεια θα προσπαθήσουν να τα καταφέρουν και ίσως χρειάζεται να τους δοθεί μια υποστήριξη έστω σε επίπεδο τεχνικό, τεχνικής υποστήριξης, όπως μπορούμε εμείς να την προσφέρουμε είτε ατομικά είτε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικώς πιστεύω ότι αν δεν καταπολεμηθεί όμως η διαφθορά, εάν δεν περιοριστεί ο, η επιρροή που μπορούν να ασκήσουν οι ολιγάρχες, δεν θα αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση στην Ουκρανία. Και φαίνεται ανεπίτευκτο, δεδομένου ότι ε, ο πρόεδρος, έχοντας μάλιστα υποστήριξη ο προηγούμενος, όντας ο ίδιος λίγο πολύ ο λιγάρχης. Ίσως, ίσως, αν και φέρεται ανεπίτευκτο κάποια στιγμή και οι ολιγάρχες οι ίδιοι να σκεφτούν ότι να, για το συμφέρον της ε, πατρίδας τους θα πρέπει να αλλάξουν συμπεριφορά. Πριν από μερικά χρόνια είχα αναλάβει μια έκθεση για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση διαφθορά στην Ουκρανία να συντάξω. Έκθεση η οποία μάλιστα προσέφερε πολύ συγκεκριμένε προτάσεις ε, για αλλαγέ και στο πολιτικό σύστημα, το νομοθετικό πλαίσιο, διάφορα θέματα δραστηριοτήτων ε, της πολιτείας, της κυβέρνησης Μάλιστα το είχαμε καταθέσει τον κύριο Παρουσένκο και τις προηγούμενες κυβερνήσεις της Ουκρανίας που όμως αγνόησαν το κείμενο αυτό, την έκθεση αυτή, όλος διόλου. Παρ' όλα αυτά εγώ θεωρώ ότι 95% τουλάχιστον αυτών των συστάσεων είναι ακόμη επίκαιρες. Μπορώ να τις καταθέσω στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή μας, εάν σας ενδιαφέρουν για να τις ε, συμπεριλάβουμε στην έκφραση υποστήριξη, στη νέα, ως έκφραση υποστήριξη στη νέα κυβέρνηση και αυτό θα μπορούσε να είναι και ένα ε, είδος δοκιμής εάν είναι διατεθειμένοι να ακολουθήσουν τις συστάσεις αυτές ε, για να καταπολεμήσουν τη διαφθορά, θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε ένα θετικό σημάδι. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τέρτς. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την Ουκρανία για τις εκλογές αυτές που ήταν άψογες σε ό,τι αφορά τις συνθήκες τις οποίες διεξήχθησαν και πραγματικά πρέπει να τους συγχαρούμε. Η αποτυχία του προηγούμενου Προέδρου στις εκλογές αυτές δεν σημαίνει ότι δεν σημειώθηκε πρόοδος στην Ουκρανία αυτά τα χρόνια η Ουκρανία ενώ ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με έδαφος της υποκατοχή μπόρεσε να σημειώσει πρόοδο. Βεβαίως πολλά πράγματα δεν προχώρησαν αρκετά γρήγορα, υπάρχουν προβλήματα με τις μειονότητες, μειονότητες υπάρχουν προβλήματα ε, λόγω τόσων ετών σοβιετικής ε, επιρροής και δεν μπορούσαν να προοδεύσουν, όμως προοδεύσαν χώρες της Δυτικής Ευρώπης στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η Πολωνία είναι 30 χρόνια, τους χάρη τώρα που οργάνωσε δημοκρατικές εκλογές. Στην Ουκρανία βελτιώνουν τα πράγματα σιγά σιγά, παρά τις δυσκολίες. Πρέπει να γνωρίσουμε βεβαίως ότι η πολιτική των Αμερικανών ίσως τελικά να είναι πιο αποτελεσματική από την Ευρωπαϊκή το soft power της Ευρώπης ήταν λιγότερο αποτελεσματικό απέναντι στους ολιγάρχες από ότι η σκληρή προσέγγιση των Αμερικανών. Και αυτό ε, είναι θετικό για την Ουκρανία. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Εμείς ε, ήμασταν πάντα ε, πολύ πιο διστακτικοί, πολύ πιο δειλοί αν θέλετε ε, απέναντι στη Ρωσία. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πιο ε, σκληροί απέναντι στον Πούτιν, διότι βλέπουμε ότι η Ουκρανία με τόσες δυσκολίες, με πόλεμο, με κατοχή, ε, δεν μπόρεσε να... Δεν, δεν, δεν οδήγησε αυτό σε στρατιωτικές λύσεις στην Ουκρανία, δεν οδήγησε σε ε, επιβολή των ολιγαρχών ε, που δεν ψήφισαν κάποιον δικό τους άνθρωπο, όχι, άλλαξε η κυβέρνηση με βάση τη λαϊκή εντολή διότι ο κόσμος όντως είχε βαρεθεί. Ε, αυτό είναι η απόδειξη ότι η ίδια η κοινωνία της Ουκρανίας είναι αυτή που επιλέγει ποιος την κυβερνάει. Και αυτή η νέα κυβέρνηση λοιπόν έχει λάβει αυτή την εντολή και θα πρέπει από πλευρά τη Ευρωπαϊκή να υπάρξει υποστήριξη. Υποστήριξη ε, πιο στεναρή έτσι, και πιο ενθουσιώδης από ότι στο παρελθόν για να ακολουθήσει η κυβέρνηση αυτή αυτό το δύσκολο δρόμο ε, που συχνά οδηγεί σε απογοητεύσεις αλλά είναι ο μόνος δρόμος για να αποδείξουμε ότι σε ένα, μια πρώην, σε σοβιετικό έδαφος μπορεί να ανθίσει μια δημοκρατία ε, που να ε, είναι έντιμη και πολιτικά και ε, διανοητικά. Φτάνουμε στους τρεις λεπτούς ομιλητές, με το που περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ο, Μίχαλ Γκάλερ, ο οποίος έχει συχνά, συχνά ήταν για την Ουκρανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία παρατηρητών και που μας μετέφεραν εδώ την εικόνα που σχημάτισαν. Νομίζω ότι συγκριτικά οι εκλογές ήταν καλύτερες από τις προηγούμενες. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αν και εγώ θα ε, ευχόμουν ότι ε, θα είχε μεταρρυθμιστεί ο εκλογικός νόμος πριν από τις εκλογές ε, γιατί νομίζω ότι το καθεστώς που επικρατεί στην εκλογική νομοθεσία δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας. Πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι το νέο αυτό κοινοβούλιο έχει 80% νέα μέλη Γι' αυτό και θέλω να σας δώσω κάποιες πρώτες εικόνες από τις πρώτες ημέρες. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει μια δημοκρατική ε, διάταξη των εδρών. Γιατί μπροστά μπροστά κάθονται όλοι οι κυβερνητικοί βουλευτέ και όλοι οι αντιπολιτευόμενοι ε, βουλευτέ κάθονται πίσω-πίσω. Δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα δημοκρατικό αυτό. Και, και εμεί εδώ στο κοινοβούλιο μα έχουμε αυτόν τον τρόπο διάταξη των εδρών, όπου τουλάχιστον ένα-δύο από κάθε πολιτική ομάδα βρίσκονται στην πρώτη θέση. Τέλο πάντων, μπορεί να είναι και λίγο οπτική αυτή η παρατήρησή μου. Αυτό που φοβάμαι κυρίω είναι ότι υπάρχει ένα κίνδυνο να ε, υπάρξει μια υπερβολική επιτάχυνση των νομοσχεδίων, της, κατα... κατάθεσης των νομοσχεδίων. Θα υπάρξει μια πλημμύρα νέων ε, νομοσχεδίων. Υπάρχουν ήδη εκατοντάδες προτάσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και βουλευτών που είναι σχεδόν αποκλειστικά άνθρωποι χωρίς κυβερνητική ή κοινοβουλευτική, ε, κοινοβουλευτική ή κυβερνητική εμπειρία. Φοβάμαι από πού ακριβώς έχουν προέλθει όλες αυτές οι προτάσεις. Έγιναν έπειτα από ε, συζήτηση σε βάθος όλων των θεμάτων που απασχολούν την ε, χώρα απο συζητηση πλαίσιο των δικών μας προσπαθειών για τη μεταρρύθμιση της ε, χώρας και των, της, μεταρρύθμισης, της μεταρρύθμισης ε, λειτουργίας του Ουκρανικού Κοινοβουλίου άλλα ελπίζαμε ότι θα συνέβαιναν. Έχουμε πλέον ένα κοινοβούλιο με ένα ε, κυβερνητικό κόμμα το οποίο έχει ισχυρή ε, πλειοψηφία. Φοβούμε μη γίνει το κοινοβούλιο ένα κοινοβούλιο σφραγίδα το οποίο απλά θα περνάει τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Μερικές φορές αυτό είναι και καλό, αλλά σε μια δημοκρατική, έφτακτη χώρα ε, νομίζω ότι αυτό δεν είναι πάντοτε θετικό. Εμείς πρέπει να, να επικεντρωθούμε στην ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα οι μεταρρυθμίσεις αποκέντρωσης, που εν μέρη έχουν ε, ολοκληρωθεί και με επιτυχία, αλλά και όλες οι άλλες μεταρρυθμίσεις. Και μια τελευταία λέξη. Αν δημιουργείται εδώ ε, η εντύπωση ότι είχαμε κάποτε υποστηρίξει ε, τον Ποροσέγκο, πρέπει να πω ότι εμείς είχαμε υποστηρίξει την κυβέρνηση που είχε ε, εκλεγεί από τον Ουκρανικό λαό. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτή την κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για πρόσωπα, μιλάμε για τον θεσμό τον οποίο υποστηρίζουμε. Και φυσικά ναι, ήταν διαφορετικό πράγμα το να συνεργάζεται κανείς με τον Γιαννούκοβιτ ή με τον Ποροσέγκο. Ξέρουμε πολύ καλά ποιο προώθησε επιτυχώ τι μεταρρυθμίσει, ποιο πραγματικά είχε την υποστήριξη υποστήριξή μας ε, για την συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα. Ευχαριστώ. Κύριος Γκέγγεση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν σήμερα εδώ για τη σημασία της υποστήριξης ε, της Ουκρανίας και της ε, βοήθειας που πρέπει να παράσουμε για να αναπτύξουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί στην Ουκρανία και να ενισχύσουν την δημοκρατική διαδικασία, τις δημοκρατικές διαδικασίες. Ε, με απότερο σκοπό βεβαίως την ενσωμάτωση της χώρας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ καλό και πρέπει να βοηθήσουμε την ε, χώρα αυτή σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση που αντιμετωπίζει. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια διάσταση την οποία δεν αναδείξαμε επαρκώς και νομίζω ε, η κυρία Μπότσκορ, η συμπατριώτησά μου, αναφέρθηκε ήδη σε κάποιες από τις ανομαλίες που αφορούν τις εθνικές μειονότητες που ζουν στην επικράτεια της Ουκρανίας. Εκείνη μίλησε για τις παρατυπίες ε, στην εκλογική διαδικασία και υπάρχουν και κάποιες άλλες παρατυπίες που εμείς οι Ούγγροι, καθώς υπάρχει ουγγρική μειονότητα στην Ουκρανία, είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Κάποιες ε, ανομαλίες που ε, αφορούν τις, τις μειονότητες στην Ουκρανία Ιδίω όσον αφορά το, την ομοθεσία για την εκπαίδευση που ε, εγκρίθηκε πριν, λίγο πριν από τις εκλογέ από την κυβέρνηση Ποροσέγκο καθώ και την ομοθεσία που αφορά τη γλώσσα. Πρόκειται για δύο νόμους που, ε, οποίους ασκήθηκε κριτική και από την Επιτροπή της Βενετίας και ε, ε, είναι θετικό το γεγονός ότι ο κ. Ζελένσκι έχει με κάποιον τρόπο, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, από άποψη ρητορική που ακολουθείται ε, τροποποιήσει τι πολιτικέ που είχαν εγκριθεί από την κυβέρνηση Ποροσέγκο. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ε, μιλά για αξίες ως προϋπόθεση για να ε, προσχωρήσει μια χώρα στους κόλπους της, να το ξεκαθαρίσουμε απόλυτα ότι τέτοιοι νόμοι είναι πέρα για πέρα απαράδεκτοι. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ε, τις δυσκολίες που έχει η οικοδόμηση έθνους και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ουκρανία, αλλά αυτά δεν μπορούν να γίνουν πρόσχημα ε, ώστε να γίνονται επιθέσεις ε, εναντίον μειονοτήτων σε πολυεθνικές χώρες. Και πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι τέτοιε τέτοιοι νόμοι είναι απαράδεικτοι. Νόμοι που στερούν ε, τις μειονότητες, ε, από τις μειονότητες τα δικαιώματά τους. Και δεν είναι μόνο τα ατομικά δικαιώματα, είναι και τα συλλογικά δικαιώματα των μειονοτήτων που πρέπει να γίνουν σεβαστά. Και ελπίζω η κυβέρνηση Ζελένσκι ε, να κάνει καλύτερη δουλειά και να διανύσει μια πιο θετική πορεία από τους προκατόχους της. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παζέσκου ο τελευταίος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι στο δυνατόν συντομότερος. Καταρχάς, όσον αφορά τη δράση της Μόσχας στην Ουκρανία. Είναι σαφές ότι επιδιώκουν διαδικασία όπως αυτή που προσπάθησαν να αναπτύξουν στην Μολδαβία δηλαδή μια ομοσπονδιοποίηση, ομοσπονδοποίηση και πρέπει να προετοιμαστούμε μια τέτοια δράση των Ρώσων. Ήθελα δημόσια να απευθύνω αυτήν την ε, προειδοποίηση στη σημερινή συνεδρίαση. Άρα, η Ουκρανία παραμένει υπό εντονές πιέσεις από πλευράς της Μόσχας, όπως άλλωστε και η Μολδαβία αυτή τη στιγμή. γιατί πάλι πρότειναν μια διαδικασία ομοσπονδοποίησης με το περίφημο πρόγραμμα COSAC. Από την άλλη, πρέπει να επιδιώξουμε να αποτρέψουμε τον εφησυχασμό στην ε, Δύση. Βλέπουμε ότι η ε, εξελίξεις στη Δυτική Ουκρανία υπονομεύουν την ε, προοπτική της ειρήνης και το κλίμα αυτό και είτε πρόκειται για την Ουγγρική είτε για τη Ρουμανική μειονότητα ή άλλες βλέπουμε ότι τα δικαιώματά τους υπονομεύονται και παραβιάζονται. Εγώ λέω ότι δεν μπορούν τώρα να λύσουν τα προβλήματα αλλά πάντως πρέπει να περιοριστεί η πίεση σε σχέση με τις μειονότητες. Έχουν πολλά άλλα προβλήματα οι Ουκρανοί και δεν θεωρούν προτεραιότητα να λύσουν τα προβλήματα των ε, μειονοτήτων. Ας τους καλέσουμε λοιπόν να δείξουν πιο θετική στάση έναντι των μειονοτήτων στην προσεχή περίοδο σαν μια λύση που θα επιτρέψει στην Δυτική Ουκρανία να μετατραπεί σε μια ειρηνική περιοχή. Σε ένα άλλο τομέα υπονομεύεται η εξουσία της πολιτικής ηγεσία των πολιτικών δομών από τις στρατιωτικές δομές. που αμφιταλαντεύονται μεταξύ Μόσχας και Ουκρανίας, καθώς έχουν περάσει την εκπαίδευση τους στην ε, Ρωσία στο παρελθόν. Έτσι λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε την ε, κυβέρνηση να επιδιώξει να βρει μια λύση για τις στρατιωτικές δομές ώστε να τις κερδίσει στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Χώρες όπως η Πολωνία, η Ρουμανία, η Τσεχική Δημοκρατία μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο καταρχάς πέρασε η μεταρρύθμιση από τις στρατιωτικές δομές πριν ε, μετά ακολουθήσει η κοινωνία. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία αντίστροφη στην ε, Ουκρανία και μάλιστα τις στρατιωτικές δομές να προσπαθούν να εμποδίσουν την εξέλιξη της χώρας. Ένα άλλο πρόβλημα που επίσης θα ήθελα να γύρω στη σημερινή συζήτηση είναι ότι θα πρέπει ενδεχομένω να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις. Αυτό πρέπει να είναι μια ορατή ε, δυνατότητα. Η Ουκρανία δεν είναι χώρα η οποία μπορεί να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις από τη μια μέρα στην άλλη και πρέπει και εμείς να δείξουμε υπομονή και ε, προσμονή ώστε να αφήσουμε τον ε, κάθε τομέα βήμα το βήμα να προχωρήσει με τα ρυθμίσεις του, διαφορετικά κινδυνεύει να μην ακολουθήσει ο πληθυσμός και το βασικό βεβαίως είναι να κερδίσουμε την υποστήριξη των πολιτών στην, ε, στις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις ουσιαστικές και ε, εις βάθος. Ας μην είναι πολύ άριθμες. Επίσης, το περιορισμένο δυναμικό της, του, του διοικητικού μηχανισμού στην Ουκρανία, γιατί ό,τι μεταρρυθμίσεις και να κάνουν δεν υπάρχει επαρκή διοικητικός μηχανισμός για να απορροφήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι, ευχαριστώ, ε, σας ευχαριστώ όλους. Θα έχουμε την Ουκρανία πολλές φορές στη συζήτησή μας. Στις 4 ε, και 4 θα έχουμε τον, την ακρόαση του νέου εκπροσώπου στο Κίεβο σε μια εντός αγωγικών ακρόαση, ας το πω έτσι. Επομένω, καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα που σας ενδιαφέρουν και επανερχόμενος προς την κυρία Καρνιέτε ε, θα επισημάνω πως βεβαίως είναι δική μας ε, επιλογή να ζητήσουμε από την ε, είπατε εκπρόσωπο να δείξει μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να δραστηριοποιηθεί στο, στο, στο θέμα της Ουκρανίας και αυτό μπορούμε να το πράξουμε με την ευκαιρία αυτής της ακρόασης. Γι' αυτό σας καλώ να είστε όλοι παρόντες. Ο κύριος Βασκόφσκι τώρα θα αναλάβει για το επόμενο θέμα να ηγηθεί, να προεδρεύσει των εργασιών.